Νομικών Θεμάτων επαλήθευσε, παρακαλώ συνάδελφε, επαλήθευσε λέγω ε, τα διαπιστευτήρια των κυρίων Πέινε, Μομπαρίκ, Πόπα, Αντέμοφ, Γιαρόκα και Πάλμερ και προτείνει να ε, ε, επικυρωθεί η εντολή τους με τι αντίστοιχε ημερομηνίε 5 Σεπτεμβρίου, 8 Σεπτεμβρίου, 13 Σεπτεμβρίου, 14 Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Υπάρχουν σχόλια? Όχι.